Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχουμε απαρτία. Όμως έχουμε το ένα δέκατο των μελών της ε, Επιτροπής. Δεν είναι σομερής ποσόστοση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αρκετούς για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ που περιμένατε όσοι ήρθατε στην ώρα σας. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν τώρα προβλέπει το σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη που είναι η παρουσίαση μιας μελέτης που έκανε ο κύριος Ζων Φρανσουά Λεμπραν. Α, όχι. Διορθώνει πρόεδρος. Θα τη την έκθεση αυτός. Αλλά είναι ένας εξωτερικός σύμβουλος που εκπώνησε την έκθεση από την Οξφόρδη. Η μελέτη αυτή λοιπόν έχει να κάνει με την οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, επιπτώσεις στην απασχόληση και τις δεξιότητες. Παρασίαση της πρόσφατης ανάλυσης 18 τομέων. Τα έχετε και στη διάθεσή σας. Δεν λέω να διαβάζετε την ώρα που θα γίνεται η παρουσίαση βέβαια. Τα έχετε όμως. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ζων Φρανσουά Ντεμπρά, καταρχήν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μας παρουσιάσει αυτή τη μελέτη και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκρόμερ. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο κύριε Λαμπρά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μίλλερ για να σας παρουσιάσει τη σύνθεση για τους 18 τομείς, θα κάνω εγώ μερικά εισαγωγικά σχόλια. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε με στόχο να ευνοήσει την προσαρμογή στις αλλαγές. Ξεκινήσαμε δηλαδή από την υπόθεση ότι αν μπορούμε να προετοιμάσουμε τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα. Δηλαδή να προετοιμαστούμε όσον αφορά την κατάθεση, την οικονομική ανάπτυξη κλπ. Και ότι θα μπορούσαμε έτσι να βοηθήσουμε με την προετοιμασία αυτή ε, την εκπόνηση και κάποιων δικτών που θα ήταν ίσως χρήσιμη για το μέλλον. Στόχος λοιπόν της μελέτης αυτής ήταν και να αναπτύξουμε κάποια νοτροπία ε, πρόβλεψης των δεδομένων και η χρήση του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και θέλαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερους φορείς και να συμμετέχουμε σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία που ήταν εκείνη των νέων προσόντων για νέες θέσεις απασχόλησης. Στόχος της μελέτης δεν ήταν ακριβώς να κάνουμε εμείς προβλέψεις, αλλά να έχουμε μια προοπτική μπροστά μας, να προβλέψουμε δηλαδή πολλά διαφορετικά σενάρια. Δουλέψαμε λοιπόν με μια μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει πολλά στάδια. Πρώτα απ' όλα ένα στάδιο το οποίο έχει ως στόχο να παρουσιάσουμε την ε, σημερινή και μελλοντική κατάσταση τομείς δραστηριότητας. Επίσης, θελήσαμε να δώσουμε κάποιες ενδείξεις για τις πιθανές εξελίξεις που θα είχαμε. Αυτά τα διαφορετικά σενάρια που σας είπα, ποιοι είναι οι παράγοντες επίσης που θα επηρεάσουν ε, την εξέλιξη. Και τέλος να δούμε τα προσόντα και τις δεξιότητες. Οι μελέτες αυτές έγιναν από ένα σύνολο εμπειρογνωμόνων ο καθένας ανέλαβε ένα συγκεκριμένο αριθμό τομέων και ανέλησε. Μας βοήθησαν βέβαια και συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Επιχείρησης. Θα σας πω δύο πράγματα και για το χρονοδιάγραμμα, γιατί θα δείτε ότι συμπεριλαμβάνεται και το Κοινοβούλιο. Τον Ιούνιο του 2006 οργανώσαμε μια μεγάλη διάσκεψη για την αναδιάρθρωση και την πολιτική ανατομέα. Και καταλήξαμε από τη διάσκεψη αυτή ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναλύσουμε τη διάσταση αυτή του κάθε τομέα. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια συγχωνεύσαμε ε, κονδύλια τα οποία μας ε, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ανάλυση για τις θέσεις απασχόλησης με κονδύλια από έναν άλλο τομέα για τις μελέτες προπτικής. Αναπτύξαμε λοιπόν μία μεθοδολογία κοινή και ξεκινήσαμε μια πειραματική μελέτη τον Οκτώβριο του 2007 για την αυτοκινητοβιομηχανία και το 2008 ξεκινήσαμε το σύνολο των μελετών. Η κάθε μελέτη, και είναι σημαντικό εδώ να το τονίσουμε, αποτέλεσε αντικείμενο συναντήσεων με εμπειρογνώμονε προκειμένου να σχολιάσουν και εκείνοι και να μας επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα. Και από τον Ιούνιο που μας πέρασε τα αποτελέσματα υπάρχουν και σε μία εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, οργανώνουμε μία μεγάλη διάσκεψη για να παρουσιάσουμε τις ε, μελέτες αυτές και να τις συζητήσουμε. Έτσι λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε και εμείς ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν για να καταλάβουμε τον ε, μηχανισμό των μελετών αυτών ότι πολλοί φορεί συμμετείχαν σε αυτές τις 18 διαφορετικές μελέτες για 18 διαφορετικούς τομείς. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όχι μόνο με τα κονδύλια τα οποία μας παραχώρησε, αλλά και η γραμματεία μας βοήθησε και συμμετείχε στις διάφορες συνεδριάσεις. Επίσης, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή Περιφερειών και η κοινωνική Εταίρη από τον κάθε κλάδο από αυτούς τους 18, το Ίδρυμα του Δουβλίνου, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και διάφορες επίσης υπηρεσίες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Έτσι λοιπόν, στο τέλος της κάθε μελέτης κάναμε εργαστήρια με ειδικού, με καθηγητές, ε, με άτομα και από άλλους ορίζοντες που ήρθαν να βοηθήσουν. Όλα αυτά σας τα λέω για να πω ότι τα αποτελέσματα θα κυκλοφορήσουν ευρέως την επόμενη εβδομάδα με το φόρουμ που θα έχουμε, αλλά θα τα παρουσιάσουμε και στις διάφορες επιτροπές ε, διαλόγου με τους διάφορους κλάδους και θα κάνουμε και δύο πράγματα επίσης ακόμα. Μία εγκάρσια μελέτη για όλους τους τομεί, για να δούμε πώ τελικά οι αρμοδιότητες, μάλλον συγγνώμη, τα προσόντα, οι δεξιότητες που εντοπίζουμε ε, σημαντικές για ένα τομέα μπορούν να χρησιμεύσουν και σε έναν άλλο τομέα. Επίσης θα αναπτύξουμε και δίκτυα, ε, παρατηρητήρια. Ε, θα φροντίσουμε να τα βάλουμε σε επαφές μεταξύ τους για να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα των προσόντων και των ε, δεξιοτήτων. Και το τελευταίο δεν θα το σχολιάσω. Είναι ένα πίνακα με τις διάφορες δραστηριότητες, τους διάφορους κλάδους για τους οποίους κάναμε ε, μελέτες. Έχουμε και νέα σχέδια, νέα προγράμματα που ξεκινάνε. Και εδώ δύο θέλω να σας πω. Είναι η εκπόνηση ενό οδηγού βέλτιστων πρακτικών για όλου αυτούς του τομείς που περνάνε από αναδιάρθρωση σήμερα. Και όπως επίσης κάτι για τη σύνδεση των δικτύων, στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, λίγα λόγια ω εισαγωγή. Ευχαριστούμε ο κύριος Μίλλερ τώρα για να παρουσιάσει την μελέτη αυτή καθ' Ευχαριστώ πολύ. Ε, την πρώτη διαφάνεια παρακαλώ. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι είναι μια πολύ εμπαριστατωμένη μελέτη, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένα πλήρη στοιχεία από εκατοντάδες εμπειρογνώμενες εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς. Και είναι, πιστεύω, μία από τις πιο πλήρεις ασκήσεις, μελέτες που έχουμε κάνει για την ανάπτυξη της, και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας. Οι τομεακές μελέτες βασίζονται σε παραδοσιακούς τομέας όπως ξυλουργικές εργασίες μέχρι τις πιο ε, προηγμένες όπως υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά, κομπιούτερς κλπ. κατασκευές. Καλύπτουμε πάνω από 60% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή ή 19 τομείς. Και έτσι σε αυτά τα δεδομένα βασίσαμε τις προβλέψεις μας. Είναι λοιπόν μια εμπεριστατωμένη ποσοτική και ποιοτική μελέτη. Όταν αναφερόμαστε τώρα στους διάφορους τομείς αυτής της παρουσίασης, αναφερόμαστε στην καρδιά, στον πυρήνα του τομέα, δηλαδή στην φάση ε, κατασκευής και συναρμολόγησης ε, αυτοκινήτων π.χ. Έχουμε μελετήσει και όλες τις διασυνδέσεις του πυρήνα με τους παράπλευρους τομείς και έτσι τα στοιχεία τα οποία θα δείτε είναι οι συγκερασμένες ε, αυτές μελέτες ή τα, τα συγκεντρωτικά στοιχεία. Αφορούν δηλαδή τον πυρήνα του τομέα σε ορισμένους τομείς όπως οι υπηρεσίες καθαρισμού έχουν βεβαίως λιγότερες διασυνδέσεις εισρωών και εκροών προς την, ε, ε, με τον επιχειρησιακό τομέα ενώ άλλες, άλλοι τομείς όπως ο κατασκευαστικός έχουν πάρα πολλές εισρωές και εκροές. Ε, θα ήθελα να τονίσω ότι εξετάζουμε και διάφορες, διάφορους τομείς σε εξέλιξη, διάφορα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα τα συζητήσουμε Δευτέρα Τρίτη στο Φόρουμ για τις Δεξιότητες ε, όπου ε, και θα οργανώσουμε και έναν αριθμό σεμιναρίων Ας δούμε λοιπόν καταρχάς ε, το βασικό ζήτημα που αντιμετωπίσαμε σε όλες τις τομεακές μελέτες Εάν δηλαδή διαπιστώνουμε εδώ μία αναβάθμιση ή μία, ένα περιορισμό υποβάθμιση των δεξιοτήτων ανατομέα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και είναι εύλογο είναι να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ υψηλών, μεσαίων και χαμηλών δεξιοτήτων και να δούμε σε ποιους τομείς αναφέρονται ποιες τάσεις. Ε, ας πούμε ότι οι υψηλών ε, δεξιοτήτων είναι η τεχνολογία ηλεκτρονικών computers, ε, στις μεσές είναι αυτοκινητοβιομηχανία, άμυνα, ε, τηλεφωνικές ε, και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και στα χαμηλά είναι οι ναυπηγοεπισκευαστικές, μη μεταλλικές εργασίες κλπ. Από απόψεως ιστορικής τώρα, όταν βλέπετε, εξετάζετε αυτούς τους 19 τομείς, όπου σας είπα καλύπτουν πάνω από, λίγο πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής απασχόλησης, ε, έχουμε ένα πολύ σαφή, μια πολύ σαφή τάση που σημειώνεται. Νομίζω στο παρελθόν δεν το είχαμε δει τόσο ε, σαφώς. Αυτό που βλέπουμε είναι μια τάση ακραία, μια τάση πόλωσης. Δηλαδή, ε, η πολύ μεγάλη ζήτηση, ψηλή ζήτηση για τις ε, δεξιότητες υψηλών προσόντων και μια δραματική μείωση της ζήτησης ε, για τα, χαμηλ, τα, τις εργασίες χαμηλών δεξιοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν βάσει αυτού του εντυπωσιακού διαγράμματος να συμπεράνω ότι αυτή η πόλωση μεταξύ ψηλών και χαμηλών δεξιοτήτων υπάρχει και επιταχύνθηκε μάλιστα τώρα στην οικονομική κρίση. Βλέπουμε λοιπόν μια επιτάχυνση της πόλωσης. Και θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε έναν άλλο σημαντικό στοιχείο, τομεακό, δηλαδή ε, τις δημογραφικές αλλαγές. Εδώ και πάλι, ε, το, το έχουμε δει και στο παρελθόν, η, το εργατικό δυναμικό γυράσκει Και μάλιστα σήμερα είναι μια επαιτειακή χρονιά, μια χρονιά όπου οι εισερχόμενοι, ο ρυθμός των εισερχόμενων είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό των εξερχομένων. Από εδώ και πέρα περισσότεροι θα εξέρχονται από, από τι θα εισέρχονται. Σήμερα έχουμε λοιπόν μια σχεδόν ισόρροπη κατάσταση, αλλά προβλέποντας τι θα γίνει στο μέλλον, προβλέπουμε πολιτική, πολιτικές τάσεις. Ορισμένες ε, διατομεακές, ε, ορισμένα διατομεακά στοιχεία. Εδώ συγκρίνουμε τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης εργασίας και ε, τις βραχυπρόθεσμες λειτουργίες έχουμε έναν αριθμό τομέων που είναι οι παραμένοντες, οι σταθεροί τομείς. Είναι βασικά οι τομείς υπηρεσιών, υψηλή αύξηση εργατικού δυναμικού, ε, χαμηλό βαθμό εξαγωγής εργασιών σε τρίτες χώρες, αρκετά ε, μεγάλο ποσοστό χαμηλών δεξιετήτων και χειρονακτικών εργασιών και η τάση που προβλέπεται εδώ ε, είναι στάσεις ε, σταθεροποιητικές ή στάσεις που δεν θα σημειώσουν, ε, θέσεις που δεν θα σημειώσουν μεγάλες αλλαγές. Εν συνεχεία έχουμε τους τομείς που αλλάζουν. Τους τομείς υπό αλλαγή που είναι βασικά οι η παραγωγή είναι, έχει, δεν έχει ανάπτυξη της, της αγοράς εργασίας, έχει μεγάλη διαφυγή εργασιών προς άλλες χώρες, ε, αύξηση των ε, θέσεων εργασίας με υψηλά προσόντα και σημαντική μείωση ε, των ειδικευμένων εργασιών και τρίτη κατηγορία είναι μετακινούμενοι τομής ε, της παραγωγής πάλι, υψηλή μείωση των, της απασχόλησης, υψηλά επίπεδα εξαγωγής εργασιών προς άλλες χώρες, το offshoring και μείωση των ε, εργασιών υψηλών προσόντων, υψηλών δεξιοτήτων. Συνολικά για σε αυτούς τους 19 τομείς κάναμε μια σύγκρουση της ετήσιας αύξησης εργασίας και της τάσης που παρουσιάζεται στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Σε πολλούς δεξιότητες, κατασκευή, ε, διατροφή, catering, έχουμε ε, αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά χαμηλά προσόντα, είναι ένας τομέας εντάσσεως υπηρεσιών. Ένα άλλο γκρουπ των εργασιών που έχουν με, μεσαίους δείκτες είναι οι τομείς εντάσσεως γνώσεων, computers, ηλεκτρονική τεχνολογία. Και η τρίτη κατηγορία είναι εντάσσεως γνώσεων και παραγωγής και εκεί είναι οι τομείς που παρουσιάζουν κινητικότητα και θα αυξηθεί το offshoring, δηλαδή η διαφυγή ε, εργασία, εργασιών σε τρίτες χώρες στο μέλλον. Ε, σε ε, μετά συνεχεία για τους 19 τομείς ε, συγκρίναμε τα μορφωτικά επίπεδα ε, όσον αφορά την δευτεροβάσμια ή τριτοβάσμια εκπαίδευση. Βλέπουμε λοιπόν έναν αριθμό τομέων όπου χρειάζονται υψηλές, υψηλά προσόντα μορφωτικά, ε, άλλους τομείς που έχουν ε, μεσαίες απαιτήσει και τρίτη κατηγορία που παρουσιάζει μια μεγάλη αύξηση του, της ζήτησης εργασίας. Τώρα, ποιοι τομείς έχουν, υφίστανται τις περισσότερες επιπτώσεις από το τρέχον οικονομικό κλίμα, την, την οικονομική κρίση. Εδώ βλέπετε με σκούρο κόκκινο, με τις σκούρες κόκκινες κουκίδες, είναι οι τομείς που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας ή που έχουν υποχρεωθεί να αναδιαστρωθούν. Παραδείγματο χάρη στην αυτοκινητοβιομηχανία υψηλέ απώλειε θέσεων εργασία και υψηλό βαθμό αναδιάρθρωση. Ο, πιο ο που θίγει πιο πολύ από όλου είναι αυτοκινητοβιομηχανία, ε, κατασκευή, χρηματοπιστωτικές εργασίες, ε, ξενοδοχειακά catering, υφαντουργία και μεταφορές. Υπάρχουν και τομείς που έχουν υποστεί λιγότερες πιέσεις λόγω της κρίσης που είναι η άμυνα. Αυτό βέβαια μπορεί να μην διαρκέσει ε, ε, μόνιμα, μπορεί να αλλάξει η ενέργεια, η υγεία και οι κοινωνικές εργασίες και η ε, ταχυδρομεία και οι τηλεπικοινωνίες. Σε αυτό το γράφημα βλέπετε την, το δίκτυ απασχόλησης. Φαίνεται περίπου λόγω θα σας εξηγήσω τι είναι. Έχουμε ε, τις ε, γραμμές, ε, τις συνεχείς γραμμές που είναι οι ιστορικές τάσεις στην αγορά εργασίας με την εξέλιξη κατά τη διάρκεια των ετών μέχρι ότου φτάνουμε στην οικονομική κρίση μετά το 2007 και μετά έχουμε κάνει προβλέψεις όχι απόλυτα επιστημονικά αλλά έχουμε υποθέσει ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται το δεύτερο εξάμεινο του χρόνου. Οι προβλέψεις βασίζονται στο σενάριο στο οποίο αναφέρθηκε ο Ζαν Φρανσουά στην αρχή. Βλέπετε λοιπόν εδώ σαφώς ότι βλέπετε τους τομείς που εφήγησαν ιδιαίτερα κατά την κρίση και ακόμα μετά από την κρίση που θα συνεχίσουν να αισθάνονται τις επιπτώσεις. Και η άμυνα έχει χάσει αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ξανακερδίσει μετά την κρίση και βλέπουμε τυπογραφικές εργασίες ε, και άλλου τέτοιου είδους υπηρεσίες να μην έχουν σημειώσει σημαντικές απώλειες. Αλλά εάν ε, ομαδοποιήσουμε τους τομείς διαφορετικά, αλλά δουν τα πράγματα. Βλέπουμε ότι στους το, παραγωγικούς τομείς ε, έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίες, ενώ στους τομείς υπηρεσιών έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας και σε συνδυασμένες εργασίες υπηρεσίες παραγωγή ε, οι στάσεις είναι και πάλι ε, ε, αυξητικές. Τώρα, μας ρώτησαν ποιες είναι οι πιο μεγάλες ε, δεξιότητες, πού θα παρουσιαστούν με τις απαιτήσει όσον αφορά δεξιότητες, σε ποιους τομείς. Θα έλεγα ότι επιγόντως χρειάζεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς, τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, δηλαδή διαπολιτισμικές δεξιότητες, ε, ε, εργασία σε ομάδες, ομαδικές ικανότητες, ε, αυτοδιαχείριση του ατόμου στην εργασία και επιχειρησιακό ταλέντο και καινοτομίες. Ε, από τεχνικής ε, τώρα απόψεως, τεχνικές δεξιότητες χρειάζονται στην τεχνολογία την, την τηλεπικοινωνιακή, στις τεχνολογίες γνώσης, στην υγεία και στις, στους πράσινους τομείς. Τώρα όσον αφορά τις δεξιότητες management διαχείρισης, εδώ πάλι διαπολιτισμικές δεξιότητες, διεθνείς δεξιότητες αξιολόγησης αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο του management, διεθνείς χρηματοπιστωτικές δεξιότητες και πράσινες, ε, πράσινα ζητήματα οικολογικά και προχωρούμε. Εάν θέλουμε τώρα να διαιρέσουμε μεταξύ των ε, τομέων ποιες είναι οι πιο ζητούμενες ε, δεξιότητες, έχουμε σε όλους τους τομείς της υγείας, τους πράσινους ε, τομείς και στο management ανάγκες και ιδιαίτερα για την παραγωγή χρειάζονται δεξιότητες στο managing και στην ε, διεθνή αλυσίδα αξιών. Επίσης ε, προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα αυξηθεί, πώς θα, τι τάση θα σημειώσει η εργασιακή αύξηση και προστιθέμενη αξία ε, σε διάφορους τομείς εργασίας, προστιθέμενη αξία και αύξηση εργασίας, η τάση, αυξητική τάση εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν στους τομείς της παραγωγής η, μειώνεται η απασχόληση αλλά έχουμε μία μεσαία και υψηλότερη αύξηση προστιθέμενης αξίας. Και Τέλος, όταν δούμε το συνδυασμό των κοινών τάσεων στην ε, τομεακή εξέλιξη, βλέπουμε ότι έχουμε τομείς οι οποίοι γυράσκουν, δηλαδή τομείς όπου χρειάζεται πηγόντως αναβάθμιση και αντιμετώπιση των προκλήσεων ε, λόγω των προβλημάτων της ε, γυρασμένης του γυρασμένου εργατικού δυναμικού, ιδίως στα ξενοδοχειακά catering, Εκεί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την άλλη πρόκληση. Δεν είναι τα, τα προβλήματα τόσο πολύ συνδεδεμένα με τη γύρανση. Ας ε, καταλήξω λοιπόν ε, στα συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, το πιο προφανές συμπέρασμα είναι αυτή η πόλωση που σας είπα που παρουσιάζεται ε, στις δεξιότητες της αγοράς εργασίας το, το είχαμε προβλέψει αυτό, ερχόταν κατά πάνω μας αυτή η, πώληση, η πόλωση στις ε, εγκάρσιες ε, τομεακές ε, μελέτες. Πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε ότι υπάρχει μεγάλη μείωση στις μεσαίες εργασίες από απόψεως δεξιοτήτων, μεγάλη αύξηση των εργασιών χαμηλών δεξιοτήτων και επίσης μεγάλη μάλλον με, τριοπαθή αύξηση της υψηλές και μεγάλη αύξηση στις εργασίες πολύ υψηλών δεξιοτήτων και θα πρέπει ε, να υπολογίσουμε ότι η, η ευρωπαϊκή αριστεία στην αγορά εργασίας ε, θα δημιουργήσει την απέτηση περαιτέρω απόκτηση ε, απόκτησης δεξιοτήτων. Πάντως βλέπουμε ότι σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται αυξημένο επίπεδο κατάρτισης. Ξεκινήσαμε μελετώντας όπως είδατε ορισμένους παραδοσιακούς τομείς όπως η βιομηχανία. Αλλά αυτή η παραδοσιακή τιμής έχουν αρχίσει θα έλεγα να αδυνατίζουν, γενικά να χάνουν το βάρος που είχαν παλιότερα, να μειώνεται δηλαδή η ζήτηση και για συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων αλλά και για ειδικέ δεξιότητες. Συνδυάζονται λοιπόν οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας με νέες ικανότητες, νέες αρμοδιότητες. Τα νέα αυτά στοιχεία έχουν σχέση με την αηφορία, σε σχέση με το κλίμα, και με την διεθνοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων γύρω από το περιβάλλον και όχι μόνο. Αλλά υπάρχει όπως είπαμε και κίνδυνος να υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένους τομείς λόγω ακριβώς της αύξησης των ηλικιών που ασχολούνται και καλύπτουν τους τομείς αυτή σήμερα. Κάποιοι επίσης τομείς θα αντιμετωπίσουν προβλήματα γιατί έχουν κακή εικόνα ανάμεσα στους νέους υποψηφίους και επίσης κάποιοι τομείς έχουν και δυσκολία στο να προσελκύσουν γυναίκες Τελειώνοντας, κάνουμε ορισμένες συστάσεις για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη εξυγχρονισμού ακριβώς των λεγόμενων ΒΕΤ, δηλαδή ε, και κατάρτιση, εκπαίδευση μάλλον και κατάρτιση, ε, να, να αντιμετωπίζουμε με πολυεπιστημονικό τρόπο τις διαδικασίες επιμόρφωσης, να καταστήσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα ικανό να προσαρμοστεί στις ανάγκες ε, των, του τομέα της παραγωγής. Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας περισσότερο σε κοινωνικές ικανότητες και σε ε, πολιτιστικές ικανότητες και γνώσεις και υπάρχει πάντα ανάγκη για πιστοποίηση και ομογενοποίηση γενικά των ικανοτήτων ε, και της διαπίστωσης ικανοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο έτσι ώστε να διασφαλιστεί με τη σειρά της η κινητικότητα. Αυτό είναι απαραίτητο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εισαγωγή ε, μέσων διδασκαλίας και κατάρτισης ε, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η διαβίου κατάρτιση θα πρέπει επίσης να προωθηθεί και η δυνατότητα επανακατάρτισης όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οι συστάσεις αυτές γενικότερα περιλαμβάνουν και έρευνα και ανάπτυξη φυσικά και καινοτομία, συνεχής επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, κάτι το οποίο είναι σχετικά καινοτόμο είναι η ανάγκη βελτίωσης ορισμένων, ε, της εικόνας ορισμένων τομέων, ιδιαίτερα για τους νέους, έτσι ώστε να καταστούν ελκυστικότερες οι δυνατότητες σταδιοδρομίας. Καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκομένους, καλύτερος διάλογος, διαφορετικές πολιτικές σχετικά με τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες, τους εκπατριστέντες ε, συστήματα παρακολούθησης της εξέλιξης ανατομία, όπως επίσης και υποστήριξη ομαδοποιήσεων και δημιουργίας δικτύων, ιδιαίτερα στον τομέα της κατάρτισης και της έρευνας και ανάπτυξης. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία θα συζηθούν στις ομάδες εργασίας που θα συνέλθουν την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ χρήσιμο, κύριε Μούλα που μας παρουσιάσατε θα έλεγα σε πρεμιέρα την εργασία αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα εργασία στον κοινωνικό τομέα. Από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει πιο αναλυτική συζήτηση, αλλά και τώρα ξεκινάει μια πρώτη συζήτηση. Η κυρία Μωρά σίγουρα θέλει το λόγο. Προς το παρόν μόνο η κυρία Μωρά θέλει το λόγο, αλλά ίσως να ανοίξει την όρεξη και σε άλλες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ακρόαση σήμερα το απόγευμα, για αυτήν την πολυτομεακή αν θέλετε παρουσίαση. Εντάσσεται στη συνέχεια αυτών που ακούσαμε σήμερα το πρωί, αλλά μας ανοίγει και συμπληρωματικές προοπτικές. Και ακριβώς τα πλαίσια αυτών των συμπληρωματικών προοπτικών να μου επιτρέψετε να επιστρέψω λίγο. Πρόκειται για μια μελέτη ιδιαίτερα τεκμηριωμένη, μια μελέτη η οποία μας επιτρέπει να δούμε κατά τομέα τις πραγματικές ανάγκες, αν και μπορεί να διαρωτηθεί κανείς αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ε, διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο μάλλον και στις διάφορες περιφέρειες στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Αλλά παρόλα αυτά κάποια σημεία συγκέντρωσαν την προσοχή μου ιδιαίτερα. Καταρχάς, η ανάγκη της λεγόμενης πολυτομεακής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξει αυτό το πράγμα περισσότερο από ό,τι σήμερα. Πρέπει να μπορούμε να συνεργαστούμε σωστά με την Επιτροπή Πολιτισμού σαν παράδειγμα για να μπορέσουμε να να πείσουμε για την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία, για περισσότερα ανοίγματα, για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και για μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυτή η πολυτομεακή δηλαδή κατάρτιση και εκπαίδευση είναι ε, τμήμα της προσπάθειας που πρέπει να κάνουμε. Το δεύτερο σημείο που προκάλεσε την προσοχή μου είναι ότι βλέπουμε ήδη να εμφανίζονται σήμερα το πρωί κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να μας απασχολήσει τα ανοίγματα δηλαδή των συστημάτων κατάρτισης και μετεκπαίδευσης στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν. Σήμερα το πρωί πολλοί εκφράσαμε τη λύπη μας στην δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι να ενταχθούν στις, ε, ε, στους χώρους εργασίας, στην αγορά εργασίας. Το άνοιγμα λοιπόν στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται των συστημάτων εκπαίδευσης είναι κομβικό σημείο και φαίνεται στην έρευνα την οποία κάνατε. Μπορείτε να με επιβεβαιώσετε αν πράγματι είναι κάτι το απαραίτητο. Και ένα τρίτο σημείο, για να μην μακρηγορήσω πρόεδρε και να δώσω και το λόγο αν ενδιαφέρεται κάποιος άλλος, θα πρέπει να βγάλουμε τα απαιτούμενα συμπεράσματα για όλες τις ανθρώπινες πλευρές αυτής της διαδικασίας. Καταρχάς, νέοι τρόποι διαχείρισης, νέοι τρόποι management δηλαδή, από τη μία και ανάπτυξη παράλληλα του, κοινωνικού διαλόγου, του κοινωνικού συγγνώμη, διαλόγου από την άλλη. Αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση και κάτι το οποίο επανέρχεται συνεχώς σε πολιτικό επίπεδο είναι αυτοί οι τρεις άξονες, πολυτομεακότητα, άνοιγμα των διαδικασιών κατάρτισης και νέοι τρόποι ε, ε, ε, ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο εργασίας μέσω των νέων τρόπων management όπως επίσης και του κοινωνικού διαλόγου. Με βάση όλα αυτά μπορούμε να βγάλουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα για τη δουλειά μας. Κύριε Μιούλερ ή κύριε Ντεμπρά θέλετε να απαντήσετε τώρα ή μετά. Ίσως τώρα να σχολιάσω για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας από τους νέους. Αν κατάλαβα καλά αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό το οποίο δείχνουν οι μελέτες οι τομεακοί είναι ένα πράγμα. Οι τομείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να προσελκύσουν νέους υπάρχουν αρκετοί λόγω της κακής εικόνας, κακές συνθήκες εργασίας κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι πολλές φορές οι νέοι ε, έχουν δυσκολία πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Απ' την άλλη αν το δούμε στατιστικά ισχύει το αντίθετο. Η αγορά εργασίας είναι αυτή η οποία δυσκολεύεται στο να προσελκύσει κάποιους νέους, τουλάχιστον σε συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις λοιπόν για αυτή την, ε, πρέπει να υπάρξουν νέες εξελίξεις για αυτή την κατηγορία ενδιαφερομένων για εργασία. Και τι πρέπει να κάνουμε πιστεύετε εσείς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Από τις τομπιακές μελέτες που έχουμε κάνει αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο ότι η απάντηση βρίσκεται στους χώρους εργασίας. Πολλά μπορεί να γίνουν λοιπόν για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας σε ορισμένες δραστηριότητες αυτό μπορεί να ξεκινήσει και από πλευρά νομοθετική. Είναι πολύτιμη η συνεισφορά του δημόσιου τομέα στο να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασία σε πολλούς τομείς. Πάντως ο ίδιο ο τομέας, οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι επιχειρήσει κτλ. πρέπει να κάνουν προσπάθειες και νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο αναγνώρισης, δηλαδή είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κυρία Φιγουερέδο. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας δώσατε, για τις μελέτες αυτές που μας είπατε. Δύο ζητήματα ουσιαστικά νομίζω ότι τίθεται τώρα. Το ένα έχει να κάνει με αυτό που είπε και χτες η Eurostat για τα ποσοστά ανεργίας. που πλήττει του νέους 20% σχεδόν. Η ανεργία πλήττει και τις γυναίκες επίσης πάρα πολύ. 10% περίπου, μέσος όρος. Η ανεργία σε ορισμένες χώρες αυξάνεται και μάλιστα με ηλικιώδεις ρυθμούς. Ιδίως στη δικιά μου τη χώρα, την Πορτογαλία. Και αυτό που μας απασχολεί είναι το εξής. Χώρες που είχαν πολύ γερούς παραγωγικούς τομείς, κυρίως τομείς όπου υπήρχε δουλειά τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους νέους, αντιμετωπίσουν σήμερα τεράστιες δυσκολίες γιατί αναδιαρθρώνονται και έτσι έχουν καταστραφεί ή μεταγκαθίστανται. Οι επιχειρήσεις κλείνουν. Συνεπώς, οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι τεράστιες. Ο παραδοσιακός κλάδος της εφαντουργίας, για παράδειγμα, στη χώρα μου, η υποδηματοπία επίσης, είναι κλάδοι που σιγά σιγά εξαφανίζονται σε περιοχές όπου ήταν ιδιαίτερα ε, παρόντες αυτοί οι κλάδοι και οδηγεί σε τεράστια ενεργεία τον πληθυσμό. Χωρίς όμως από την άλλη μεριά να έρχονται νέες θέσεις απασχόλησης που να αντικαθιστούν αυτές που χάνονται. Και ας γίνονται κάποιες επενδύσεις. Οπότε η μελέτη σας υποθέτω ότι δεν λαμβάνει υπόψη αυτό το στάδιο. Και γι' αυτό έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, Κατά τη γνώμη σας, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε. Πώς είναι δυνατόν η κατάρτιση των νέων και του, των ανέργων γενικότερα Τι προπτικές υπάρχουν ώστε να φροντίσουμε να προσαρμόσουμε και την κατάρτιση τι δηλαδή προτάσεις για απασχόληση μπορούμε να έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν μιλάω τώρα για μετά από τέσσερα χρόνια, για τώρα αμέσω τι έχουμε να τους προτείνουμε. Γιατί δεν τολμάω να σκεφτώ τι θα γίνει μετά από μερικά χρόνια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος Μίλλερ να απαντήσει. Καταρχάς, σύμφωνο ε, με μια παρατήρηση του προλαλήσαντος ότι σε αυτή την παρουσίαση θεωρήσαμε την Ευρώπη ολόκληρη. Δεν κάναμε διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών και των περιφερειών. Σωστή παρατήρηση. Και συμφωνώ ότι αν είχαμε κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, η εικόνα θα ήταν διαφορετική ανάλογα με την περιφέρεια. Επίσης είναι σωστό ότι σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένους τομείς, η τρέχουσα οικονομική κρίση είχε τεράστιες επιπτώσεις. Έχει χτυπήσει πολύ άσχημα. Ιδίω στην Πορτογαλία, ορισμένοι τομεί τη βιομηχανία αποτελούν ένα καλό παράδειγμα αυτού του γεγονότο. Όταν μιλάμε για την κλωστοϊφαντουργία, εννοούμε ότι αυτή η δυσμενής κατάσταση είναι η συνέχιση μιας ε, παλιότερης κρίσης, μιας κρίσης του παρελθόντος η οποία έχει οξυνθεί λόγω της κρίσης και ε, λόγω της, των αναδιορθώσεων που έκαναν πολυεθνικές εταιρείες και άλλων γεγονότων. Η πρόκληση εδώ που αντιμετωπίζουμε είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μία ιδέα ε, για το πότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Και Βάσει των υπολογισμών που κάναμε, σας είπα ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2010 πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε να σηκώνουμε κεφάλι. Μπορεί να είναι βέβαια και αρχή του 2011. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να επιμικίνουμε την σημερινή κρίση με εσφαλμένα μέτρα τα, τα οποία θα οδηγήσουν σε μια παράταση της κατάστασης. Εάν κοιτάξετε τώρα την ανεργία των νέων, ασφαλώς δεν είναι ευχάριστα τα στοιχεία σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένους τομείς, για συγκεκριμένες ηλικιακέ ομάδες δηλαδή. στον πολύ καλή ερώτηση για το τι μπορεί λοιπόν να γίνει. Πιστεύω ότι αυτό το ερώτημα είναι το ερώτημα κλειδί το οποίο θα συζητηθεί Δευτέρα Τρίτη την ερχόμενη εβδομάδα. Η τομεακέ μελέτες ολοκληρώθηκαν περίπου πριν από ένα χρόνο. Ορισμένε από τα σεμινάρια των εμπειρογνωμών οργανώθηκαν στην αρχή, του τρέχοντος έτους αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι μόλις τότε είχαμε καταλάβει το βάθος της οικονομικής κρίσης και προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε αυτό το επιπλέον στοιχείο στις τομιακές αναλύσεις, όπως έχουν σήμερα, δεν υπάρχουν πολλές προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε πρόθεσμα, να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Είναι το ερώτημα, το κεντρικό, το ερώτημα κλειδί του φόρουμ, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα Τρίτη. Η κυρία Ντιτ Μπάουρ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, Έχω λάβει μία απάντηση σε μία ερώτησή μου ήδη, διότι εξεπλάγει όταν είδα τα γραφήματα ότι στον τομέα των κατασκευαστικό και στον τομέα των μεταφορών είναι οι λεγόμενοι τομείς οι οποίοι παραμένουν στην ίδια κατάσταση. Ενώ πολύ πρόσφατα οι οδηγοί των φορτηγών είχαν εκφράσει έντονα παράπονα για τις οδικές μεταφορές και είχαν πει ότι έχουν χάσει 50%, 50% των εργασιών τους. Εξεπλάγει λοιπόν που αυτή η τομή είναι υπό τον ε, όρο σταθερή, σταθερή στην κατηγορία σταθερή. Ίσως ε, τα προβλήματα αυτά να είχαν σημειωθεί πριν ξεσπάσει η κρίση και γι' αυτό παρουσιάζονται έτσι ως ε, σταθεροί. Σήμερα το πρωί ακούσαμε σε τα παρόμοια προβλήματα υπό διαφορετική οπτική γωνιά. Μία από τις ε, εκθέσεις που παρουσιάστηκαν το πρωί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις υψηλές, στα υψηλά προσόντα, στις υψηλές δεξιότητες της, κατασκευασ... της παραγωγής ε, και σε εξειδικευμένους εργαζόμενους. Οι σας, ε, τα δικά σας συμπεράσματα είναι διαφορετικά από την προηγούμενη μελέτη. Οι δικές ε, σας μελέτες καταλήγουν σε άλλο συμπέρασμα ότι δηλαδή η ζήτηση για αυτού του είδους χαμηλών, ε, χαμηλής κατάρτισης, χαμηλόβασμης κατάρτισης ε, μειώνεται. Πώς μπορείτε να εξηγήσετε αυτήν την αντίθεση. Μία άλλη ε, ένα άλλο συμπέρασμα που ακούσαμε το πρωί είναι ότι στην Ευρώπη οι απόφοιτοι της δευτεροβάσμιας εκπαίδευσης είναι εγκαταλείπουν τη σχολική εκπαίδευση σε υψηλά ποσοστά. Σε ορισμένε χώρε 14% δεν τελειώνουν καν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ε, μετά αφού το άκουσα τα σχόλιά σα, σκέφτηκα ότι αυτά τα άτομα, αυτοί οι νέοι, οι οποίοι είναι, έχουν πάρα πολύ χαμηλά προσόντα, πολύ λίγες δεξιότητες, θα πρέπει να αναλυθούν το φαινόμενο δηλαδή αυτό, αυτή η ομάδα περισσότερο, ε, για να δούμε πώς μπορούν ε, να ενταχθούν, τι προοπτικές έχουν, δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για εργασίες και την ε, ζήτηση περισσότερων προσόντων. Επίσης, ε, θέλω να πω ότι η μελέτη αυτή ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα λάβω υπόψη όλα τα στοιχεία που αναφέρονται και θα ήθελα να έχω ένα hard copy αυτής της έκθεσης διότι ήταν πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα γραφήματα. Θα ήθελα λοιπόν να τα έχουμε στο φακέλους μας ε, την ε, μελέτη αυτή που είναι πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ. Καταρχάς αυτό που είπατε για τους τομείς που παρουσιάζουν μια σταθερότητα ε, είναι οι τομείς οι οποίοι, όπου δεν χάνονται πολλές εργασίες στο εξωτερικό σε άλλες χώρες, κατασκευή, μεταφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες, όπως η παραγωγή φορτηγών ή κατασκευαστικών υλικών, ε, δεν κατασκευάζονται αλλού. Αλλά βασικά το επίπεδο του offshoring, επειδή είναι βασικά ντόπιε οι κατασκευαστικέ αυτές βιομηχανίε και οι βιομηχανίε παραγωγής δεν σίγονται τόσο πολύ όπως άλλοι κλάδοι, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Έχουν λοιπόν χαμηλό επίπεδο offshoring. Εν, συνεχεία, συγκρίνατε ορισμένα στοιχεία από την πρωινή μελέτη την οποία εγώ δυστυχώς δεν παρακολούθησα και αν κατάλαβα καλά το πρωί το συμπέρασμα έλεγε ότι ε, προτείνεται η επιτάχυνση της απόκτησης υψηλών δεξιοτήτων στον τομέα, τον παραγωγικό κλπ. Ναι, εμείς αναφερθήκαμε στην ευρωπαϊκή αριστεία, παραγωγική αριστεία. Στη δικιά μας μελέτη έχουμε, αν θέλετε, δύο παραγωγικούς τομείς. Και στους δύο πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις υψηλές δεξιότητες Παρόλα αυτά, σε ορισμένου τέτοιου υψηλού παραγωγικού τομεί, δεν θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε την διαφυγή εργασιών, όπως είπα, στην κλαστοϊφαντουργία. Ενώ αυτές οι δεξιότητες για τις οποίες θα υπάρχει ακόμα ζήτηση στην Ευρώπη θα είναι μόνο αυτές των υψηλών προσόντων. Δεν ξέρω λοιπόν κατά ποιο βαθμό συμφωνούν τα συμπεράσματά μας με την πρωινή έξεση. Οι δικές μας μελέτες επίσης καταλήγουν στο ότι ο τομέας των υπηρεσιών και οι χαμηλών δεξιοτήτων εργασία έχουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξη εργασία. Και μετά την κρίση αυτή πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης που αντιτίθεται ε, στην τάση ότι θα αυξηθούν μόνο οι υψηλών προσόντων εργασίας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει μια μεγάλη αγορά εργασίας που ζητάει χαμηλές ε, δεξιότητες, ε, χαμηλού επίπεδου προσόντα. Όπως είπατε, πολλοί που εγκαταλείπουν το σχολείο ή τελειώνουν το σχολείο, ιδιαίτερα αγόρια, εκεί υπάρχει ψηλή ανεργία και πάντοτε στην Ευρώπη τουλάχιστον θα υπάρχει δυνατότητα απορρόφησής τους σε μια αγορά ε, ε, μεγάλη αλλά πολύ χαμηλών προσόντων. Και συνήθως ε, τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να προωθηθούν σε τομείς που όμως έχουν μια χαμηλή εικόνα κοινωνική, δηλαδή ε, δεν αξιολογούνται κοινωνικά όσο άλλοι τομείς ψηλών δεξιοτήτων και έχουν μια αρνητική εικόνα. Και τέλος, για τα ντοσιέ σας, για του φακέλους σας, η παρουσίαση μου αυτή ήταν 15 λεπτών, αυτό αυτό το όριο είχαμε, θα μπορούσα να την κάνω 50 λεπτών ή θα προσιάσω τη Δευτέρα τουλάχιστον μια ε, ομιλία 50 λεπτών, ε, μια πιο εμπεριστατωμένη ομιλία με περισσότερα στοιχεία. Και ευχαρίστως ε, να την ε, δώσω στους συναδέλφους από την Κομισιόν. Τη Δευτέρα λοιπόν θα είναι η πλήρης ομιλία, η ε, παρουσίαση της μελέτης. Εδώ ήταν λίγο συντετμημένη. Ευχαριστούμε κυρία Ράπτη. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, το πρώτο που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που είχατε να διοργανώσετε αυτή την ακρόαση με τις μελέτες, και την απογευματινή και την πρωινή. Έτσι ε, έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή μας θα μπορεί να εργαστεί πολύ καλύτερα και πολύ αποδοτικότερα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και τα πρωινά δεδομένα, όπως και τα δεδομένα της μελέτης που ακούσαμε απόψε. Ε, τρία σημεία θέλω να βάλω στην ε, κουβέντα. Το ένα σημείο έχει να κάνει με το δημόσιο άκουσα από τον ομιλητή ότι υπάρχει πάντα η προοπτική του δημόσιου τομέα. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε έντονο πρόβλημα σε σχέση με την ανεργία και σε σχέση με τη δυνατότητα να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ε, σημειώνω ότι η νέα κυβέρνηση των σοσιαλιστών έχει πάρει μία απόφαση που λέει ότι στο δημόσιο τομέα για κάθε πέντε υπαλλήλους που θα φεύγουν θα προσλαμβάνεται ένας αυτό είναι ένα αριθμητικό στοιχείο που πραγματικά θα ήθελα να δω πώς μπορεί να σχολιαστεί από την πλευρά των μελετητών. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τα προσόντα. Υπάρχουν πάντα οι θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερα προσόντα, χαμηλά προσόντα. Και εδώ θέλω να βάλω τη διάσταση της μετανάστευσης. Στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω και σε άλλες χώρες, πάρα πολλές θέσεις εργασίας που απαιτούν χαμηλά προσόντα καλύπτονται από μετανάστες. Είναι και αυτή μέρος της παραγωγικής διαδικασίας και θέλω να ρωτήσω κατά πόσον έχει μετρηθεί η συνεισφορά τους. Το τρίτο και τελευταίο σημείο έχει να κάνει με, την, με τις ηλικίε της ανεργίας. Υπάρχουν οι νέοι οι νέοι που παίρνουν πολλά προσόντα και μένουν χωρίς δουλειά, ε, και αυτό το κάνει περισσότερο οξύ το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και οι λιγότεροι νέοι, οι οποίοι είτε έχουν περισσότερα προσόντα είτε λιγότερα προσόντα, ε, χάνουν μία δουλειά σε μία ηλικία που μπορεί να είναι από 35 ως 50-52 και για αυτούς είναι ακόμα πιο δύσκολο το να βρουν εργασία ανεξάρτητα από τα προσόντα που έχουν. Πάρα πολλοί δε από αυτούς αναγκάζονται να δεχτούν μια εργασία, με πολύ λιγότερα, μια εργασία που να απαιτεί πολύ λιγότερα προσόντα από αυτά που πραγματικά έχουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το πρώτο για το δημόσιο τομέα και την ε, ανεργία. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα απόλυτα καλά το παράδειγμα που μου δώσατε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό πάντως εδώ να σημειώσουμε ότι η υγεία, οι κοινωνικές παροχές είναι πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται στη μελέτη και σίγουρα αποτελούν ένα τεράστιο τομέα που περιλαμβάνει ένα σωρό θέσεις απασχόλησης σε διάφορα επίπεδα. Η μελέτη αυτή καταλή ε, περιλαμβάνει πάνω από 20% της απασχόλησης. Ένα τεράστιο μέρος της ιδιωτικής απασχόλησης αλλά και μέρος της δημόσιας απασχόλησης. Απασχόληση στο δημόσιο δηλαδή. Όπως σας είπα, κοινωνικός τομέας, υγεία, τηλεπικοινωνίες που εν μέρη μπορεί να είναι δημόσιος τομέας. Εγώ έχω περιλάβει στη μελέτη αυτή λοιπόν όλους αυτούς τους τομείς. Τώρα, και ο κοινωνικός τομέας και η υγεία περιμένουμε ότι θα προσφέρει περισσότερες θέσεις απασχόλησης στο μέλλον. Με ρωτήσατε επίσης για τους ανθρώπους χαμηλών προσόντων και τους μετανάστες, κατά πόσο υπάρχει αξιολόγηση για την συνεισφορά τους. Η απάντηση είναι όχι δυστυχώς. Δεν έχει γίνει. Δεν αποτελεί μέρος της μελέτης μας. Υπάρχει κάποια μικρή διάσταση η οποία αναφέρεται στο πώς οι διάφοροι κλάδοι πιστεύουν ότι μπορούν να ε, λυθούν τα προβλήματα έλλειψης εργατικού δυναμικού εκεί όπου υπάρχει έλλειψη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όσον αφορά τη συνεισφορά των ε, μεταναστών, όχι, αυτό δεν καλύπτεται από, την ε, μελέτη, από τις μελέτες αυτές των διαφόρων κλάδων. Και το τελευταίο ήταν για την ηλικιακή ε, ζώνη 35 με 50. Είναι ηλικίε ακριβώς που έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αυτή η ηλικία, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Έχουν εμπειρία. Συνήθως είναι καλύτερα καταρτισμένοι έχουν εμπειρία από την αγορά εργασία αν το συγκρίνουμε με άλλες ηλικίε, βέβαια. Οπότε, η ηλικία αυτή 35 με 50 δεν έχει εντοπιστεί σαν ε, που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Θέλω να ολοκληρώσω εδώ με το εξή. Το βασικό για μας ήταν η κλάδη εδώ. Ανακλάδο εξετάσαμε το πρόβλημα. Πώς έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα, πώς αντιμετωπίζουν την κρίση και τι μπορούμε να περιμένουμε μετά την κρίση, όποτε και αν αυτή τελειώσει. Η προσέγγιση μας λοιπόν είναι λιγότερο αναχώρα ή αναπεριφέρειες ή αναομάδες εργατικού δυναμικού. Δεν ήταν αυτή η προσέγγιση μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μιλάμε για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και συνήθως υπογραμμίζουμε πόση σημασία έχει οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα προσόντα, περισσότερες ε, δεξιοτεχνίες. Και μάθαμε επίσης, ακούσαμε ότι καλό είναι να υπάρχουν πολλαπλά προσόντα. Οι δάσκαλοι τώρα, το διδακτικό προσωπικό, πώς προετοιμάζεται για αυτές τις αλλαγές που έχουμε στην αγορά εργασίας. Πώς με τη σειρά τους θα καταρτήσουν σωστά αυτούς που ζητάνε βοήθεια από αυτούς. Οι τομεϊκές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μια ανάγκη ε, ε, κατάρτισης των εκπαιδευτών, Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε πολυπολιτισμικές δεξιότητες. Ασφαλώς, λοιπόν, πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους εκπαιδευτές, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό το στοιχείο έχει περιληφθεί στις μελέτες μας. Ευχαριστώ. Έχετε να κάνετε άλλες ερωτήσεις. Μία ερώτηση. Συμπερασματικά θα έλεγα. Ξέρετε ότι έχουμε εμπλακεί στην διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα δέκα χρόνια. Και βλέποντας τα συμπεράσματα της δικής σας μελέτης, τι θα λέγατε στους πολιτικούς για το τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και να εκμεταλλευτεί πλήρως θα έλεγα αυτήν την η ιδιαίτερα αναλυτική και λεπτομερή εργασία την οποία παρουσιάσατε. Μου έκανε εντύπωση ένας πίνακας τον οποίο έχετε όπου οι μέσες ικανότητες είναι πολλές φορές δεν ζητούνται Δηλαδή δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ξέρουν μόνο να γράφουν και να διαβάζουν και να μετρούν, αλλά θα πρέπει επίσης να ομιλούν την αγγλική και να γνωρίζουν και να εργάζονται στο διαδίκτυο. Αυτές είναι οι λεγόμενες μέσες ικανότητες ενός εργαζομένου. Ε, και παρόλα αυτά δεν τις εκμεταλλεύεται η αγορά εργασίας πλήρως αυτές τις ανάγκες. Γιατί γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτοί οι αριθμοί μας ανησύχησαν και μας. Τι γίνεται ακριβώς εδώ. Το θέμα δεν είναι η ηλικία, δηλαδή 35 με 50. Είναι ουσιαστικά ο σκέλετος της κατασκευαστικής γενικότερα ε, δραστηριότητας στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το σύνολο της οικονομικής ανάπτυξης αυτή μειώνεται μέχρι τώρα και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν να παίρνετε ένα τρένο και φτάνετε στο σταθμό, ε, μία φωνή σας λέει προσέξτε το κενό με την αποβάθρα, mind the gap. Αυτό μας λέει ουσιαστικά αυτή η έρευνα, φωνάζει αυτή η έρευνα, προσέξτε το κενό. Από τη μία βλέπουμε ότι δημιουργούνται ε, πολύ περισσότερες θέσεις χαμηλών απαιτήσεων στην Ευρώπη από ό,τι περίμενα. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους νέους να εκπαιδευτούν σωστά. Παρ' όλα αυτά βέβαια υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένους τομείς και σε αυτή την κατηγορία λόγω των κακών συνθήκων εργασίας και των χαμηλών αμοιβών. Αλλά ίσως σε κάποια φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι σε θέση να απορροφήσει υποψηφίους εργαζομένους υψηλού επίπεδου. Γνωρίζουμε επίσης ότι αν έχει κανείς πανεπιστημιακό δίπλωμα, υψηλές ικανότητες κτλ. Όλα αυτά τώρα πια είναι θα έλεγα θεωρητικά. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το τι σημαίνει στη μέση των ικανοτήτων που απαιτούνται. Εκεί είναι η μεγάλη κατηγορία στην οποία αναμένεται να υπάρξει συνέχεια στη ζήτηση. Και γι' αυτό ακριβώς ε, λέμε ότι ανάμεσα στις κατώτερες θέσεις και στις ανώτερες προσέξτε το κενό. Το τι μεσολαβεί δηλαδή ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Δηλαδή εσείς θέλετε να συμπέσει το στοιχείο της ανάλυσης σας αυτό με την τομεακή σας ανάλυση. Αυτό ισχύει που λέτε για τους λεγόμενους εισαγωγικά παραδοσιακούς παραγωγικούς τομείς. ενώ ε, ίσως να μην ισχύει για τους λεγόμενους καινοτόμους τομείς. Εκεί δεν βλέπετε πάρα πολλά πράγματα να γίνονται στο εσωτερικό της Ένωσης. Δεν ξέρω αν σας καταλαβαίνω καλά. Αυτό το οποίο στοχεύεται είναι η φαντουργία, η αυτοκινητοβιομηχανία, τέτοιου είδους παραδοσιακές εισαγωγικά δραστηριότητες. Νομίζω ότι περνάμε λίγο περισσότερο και δεν περιοριζόμαστε στην υφαντουργία και στα αυτοκίνητα. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει παραγωγή στην Ευρώπη στο μέλλον, αλλά θα εξυπηρετείται κυρίως από ανθρώπους με υψηλές ικανότητες. Και οι δραστηριότητες που δεν απαιτούν υψηλές ικανότητες δεν θα γίνονται πια στην Ευρώπη. και ακριβώς θα υπάρχουν ανάγκες για ανθρώπους οι οποίοι να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν ακριβώς την καινοτομία, την έρευνα κτλ. Και όλες τις υπηρεσίες οι οποίες πηγαίνουν μαζί. Δεν λέγω ότι θα φτάσουμε σε μια υπηρεσία 100% υπηρεσιών, αλλά το παραγωγικό κομμάτι θα έχει περισσότερο σαν στόχο τους εργαζομένους με υψηλές δυνότητες απασχόλησης και όχι τόσο τους εργαζομένους του κάτω τμήματος της κλίμακας. Και η πρώτη μου ερώτηση, τι πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η βασική πρόκληση που έχουμε είναι οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και για αυτούς τους εργαζομένους. Βέβαια η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι θέλουμε καλύτερες θέσεις σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω παρόλα αυτά ότι από τη μία πλευρά του κενού θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις συνθήκες εργασίας. Από την άλλη πλευρά, στο υψηλό τμήμα, έχουμε έτσι και αλλιώς το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, έχουμε δυνατότητες ε, έρευνας και ανάπτυξης, υπάρχουν εκεί δυνατότητες. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. αλλά το θέμα των καλύτερων συνθήκων εργασίας είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει. Έχει τελειώσει ο κατάλογος των ομιλητών η κυρία Μογά. Μια ερώτηση η οποία επανέρχεται συνεχώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μήπως θα πρέπει να ε, δουλέψουμε και λίγο στις ε, αντιλήψεις που έχουμε νοητικά για συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης. Όχι μόνο στις συνθήκες της εργασίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται και βλέπουν τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Ναι, αλλά θα έλεγα Καταρχάς, να αλλάξουμε την πραγματικότητα επειδή υπάρχουν πάρα πολλές συνθήκες εργασίας που δεν είναι καλές. Όταν αλλάξουμε την πραγματικότητα, το τι ισχύει σήμερα, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Λεμπρά, από πλευράς Κομισιόν. Και εγώ εκμεταλλεύτηκα αυτή την ανταλλαγή απόψεων, αλλά. Αναρωτιέστε και εσεί, όπως και ο κύριο Μίλλερ τελικά, τι θα γίνει με αυτή τη μελέτη, πού θα πάει, αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε και εσά. Πείτε μας, τι θα γίνει με αυτή τη μελέτη, ποιο δρόμο θα πάρει. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές. Η πρώτη ανταποκρίνεται στις απορίες που έχετε όσον αφορά το μέλλον εντός αγωγικών της απασχόλησης. Όμως πρέπει πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε ότι οι μελέτες αυτές είναι μελέτες που ξεκίνησαν ως διαρθρωτικές. Αυτό ήταν ο στόχος. Δεν αναλύουν δηλαδή βραχυπρόθεσμα την ε, εξέλιξη, ούτε πρόκειται για προβλέψεις. Πρόκειται για προοπτική που δίνουν για το ποιες θα είναι οι μεγάλες προκλήσεις στους τομείς αυτούς. Άρα δεν μιλάμε για την κρίση, είμαστε πέρα από αυτό. Γιατί η κρίση είναι αλήθεια ότι επιταχύνει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτό ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όταν μιλάμε για σενάρια, για προοπτικές που δίνουμε, αυτό που κάνουμε είναι ότι μιλάμε για μελλοντικές στρατηγικές. Τι θέλουμε να πετύχουμε, πού μπορούμε να δράσουμε, γιατί κάπου αλλού δεν μπορούμε να δράσουμε. Εμείς σας δείχνουμε πού νομίζουμε ότι μπορούμε να παρέμβουμε για το αφορά τη δημογραφία, την αγοραστική δύναμη, την παγκοσμιοποίηση. Εκεί Ελάχιστα μπορούμε να επηρεάσουμε. Μπορούμε όμως να φροντίσουμε για την κατάλληλη ρύθμιση. Να αναπτυχθεί η έρευνα και η ανάπτυξη, η κατάρτιση, η εκπαίδευση. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα λοιπόν για αυτά. Για να απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Άμυνα. Να, ένα, <clears throat> ένας κλάδος που μελετήσαμε. Υπάρχει προγραμματισμός που ανταποκρίνεται στις οικονομίες κλίμακας. Ε, για την απασχόληση. Μπορούμε να φτάσουμε βέβαια σε ένα τεράστιο ανταγωνισμό. Λοιπόν, μια από τις οδούς που προτείνουμε είναι ότι δεν προσπαθούμε να ε, συμφωνήσουμε μεταξύ μας για την έρευνα, την ανάπτυξη, τις αγορές, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε καλύτεροι από τους καλύτερους και να μπορούμε να εξάγουμε. Είναι και το εμπόριο όπλων, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά είναι και αυτός ένας κλάδος που αναλύσαμε. Έρχομαι σε άλλο κλάδο, η φαντουργία. Είναι σαφές, το λέει αυτή η μελέτη αλλά και πολλές άλλες, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαζική παραγωγή με ε, συγκριτικό πλεονέκτημα. Είμαστε όμως οι καλύτεροι όσον αφορά την ποιότητα. Είτε πρόκειται για το δέρμα, είτε για το ύφασμα. Το ίδιο ισχύει και για άλλους κλάδους που έχουν να κάνουν με την υφαντουργία. Έχουμε και την κατάρτιση, όπου σήμερα βρίσκουμε περισσότερους Κινέζους Ινδούς από ότι από τις νέες ευρωπαϊκές χώρες γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης. Άρα χρειάζεται περισσότερη συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης. Για να σας πω δηλαδή ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε χωρίς να υπάρχει μία λύση θαυματουργή. Αλλά υπάρχουν πολλές επιμέρους λύσεις που όλες μαζί μπορούν να βοηθήσουν. Ο Κιμίλερ το κατέδειξε ότι υπάρχει μια αλυσίδα αξιών. Γιατί η βιομηχανία μπορεί να είναι μικρή στην απασχόληση, αλλά είναι αναγκαία για να δημιουργηθεί πλούτος. Πολλοί κλάδοι εξαρτώνται από τη δημιουργία αυτή του πλούτου και της προστιθέμενης αξίας. Και κάτι ανησυχητικό όσον αφορά την απασχόληση. Στα workshop που κάναμε με τους εμπειρογνώμονες, και αυτό το είδαμε για όλους τους κλάδους, τους ρωτήσαμε ε, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα των προσλήψεων. Ε, προσλαμβάνετε αυτή την κατηγορία ή την άλλη κατηγορία. Και μεταξύ άλλων υπήρχαν και οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Τι είπαν? Όχι. Είναι ο τελευταίος που θα πάρουμε. Θα προτιμήσουμε να πάρουμε ξένους, μετανάστες, αλλά όχι μακροχρόνιους άνεργους. Ε, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει δουλειά με στόχους μακροπρόθεσμους μερικές φορές. Να βλέπουμε και το μέλλον. Γιατί ο χρόνος είναι μια πολύ επικίνδυνη μεταβλητή. Χρειαζόμαστε χρόνο για να προετοιμαστούμε. Συγχρόνως όμως, αν περιμένουμε και δεν είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, ξαναπάρουμε αυτούς τους ανθρώπους στην αγορά εργασίας. Και σίγουρα μας απογοητεύει, γιατί είπαμε δεν μπορούμε εμείς να προβλέψουμε το μέλλον, δεν μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή διάφορες εναλλακτικέ χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι πρόβλημα θα έχουμε. Για μερικά όμως ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να έχουμε μαζική παραγωγή για το ύφασμα. Οπότε, οπότε ας ακολουθήσουμε κάποια άλλη εναλλακτική. Και κάτι ακόμα που υπογράμμισα και πριν. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους του κάθε κλάδου για να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Και κυρίως για να προσπαθήσουμε να έχουμε και τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων που έχουν λόγο σε αυτά. Στις μελέτες μας διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει αρκετή ανταλλαγή απόψεων με όλους αυτούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την ίδια ανάλυση, την ίδια προβληματική, την ίδια εξέλιξη της απασχόλησης στην εφεδεουργία, αλλά ανταλλαγή απόψεων δεν υπάρχει. Άρα και εδώ, και αυτή είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Αν θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, πρέπει να έχουμε τις δεξιοτεχνίες που χρειάζεται και μόνο τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομίες κλίμακας. Όταν ανταλλάσσουμε απόψεις και έχουμε περισσότερα κοινά ε, ιδρύματα κατάρτισης μεταξύ μας. Ευχαριστούμε. Τότε όμως πρέπει να δούμε τι έγινε με την περίπτωση του τέλο, που αντί να αλλάξουμε ένα εργοστάσιο και να το κάνουμε από μεγάλους υπολογιστές γραφείου φορητούς υπολογιστές με απολύσεις που δεν βλέπουμε πότε θα βγουν από αυτή την ε, ανεργία να σκεφτούμε καλύτερα το θέμα αυτό τη εγκατάσταση του εργοστασίου στην ε, Πολωνία. Δεν λέω ότι θέλω να το σχολιάσετε αυτό, όχι. Αλλά σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ, για τα όσα μα μάθατε και για όσα μα εξηγήσατε προκειμένου να αναλύσουμε καλύτερα την επόμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Την επόμενη φορά θα βρεθούμε 26 και 27 Ιανουαρίου. Διακόπτουμε λοιπόν. Λίγη εδώ η σημερινή μας συνεδρίαση. Όσοι συμμετέχουν όμως στην ομάδα εργασίας γυναικών να παραμείνουν παρακαλώ στην αίθουσα.